Good afternoon, dear colleagues. I invite you... Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Για να αρχίσουμε τις εργασίες μας για σήμερα το απόγευμα. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι το ψήφισμα για την ε, διάσκεψη COP23 του 2017 που θα γίνει στην ε, Βόνη, 16 Νοεμβρίου. Και πριν δώσω το λόγο στους συντάκτες του ψηφίσματος αυτού, ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, αυτής, και επειδή θα συμμετέχω στην αντιπροσωπή αυτή που θα πάει στη Βόνη, θέλω και εγώ να πω μερικά πράγματα. Ήταν πάντα μεγάλη πρόκληση να έχουμε μια συμφωνία. Το πετύχαμε στο Παρίσι, ευτυχώς, και είμαστε βέβαια ιδιαίτερα ευτυχείς με το επίτευγμα αυτό. Τώρα, με τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που έχουμε από πλευρά των ΗΠΑ, θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουμε επίση επίσης μεγάλη δυσκολία. Πώς θα τηρήσουμε δηλαδή τις υποχρεώσει που έχουμε αναλάβει σε διεθνές επίπεδο. Η γρήγορη κύρωση και θέση σε ισχύ της συμφωνίας αυτής είναι κάτι πολύ θετικό. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα για να πετύχουμε τους στόχους μας, παρόλο που αποσύρεται από ό,τι φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες από την συμφωνία αυτή. Οπότε δεν θα υπάρχει η δικιά της εθνική συγχρηματοδότηση θα πρέπει να φροντίσουμε να το καλύψουμε εμείς. Επιπλέον, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κοινοτόμα νομοθεσία να μας βοηθήσει να πετύχουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο Παρίσι. Αυτή η νομοθεσία υπάρχει, είναι το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα. Και να συνεχίσουμε και να ε, προωθήσουμε και να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Να χρησιμοποιήσουμε και τα μέσα που διαθέτουμε στα πλαίσια της διεθνούς διπλωματίας. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά που έχουμε υπογραμμίσει και στο ψήφισμά μας αυτό το κοινό. Σίγουρα, πολλοί συνάδελφοι θα έχουν να προσθέσουν διάφορα πράγματα. Εμείς λοιπόν θα συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις στη Βόνη και χωρίς άλλη καθυστέρηση. Θέλω να δώσω το λόγο στους συνυπογράφοντες. Και βέβαια και όποιος άλλος μετά θέλει το λόγο, ευχαριστώ. Πρώτος. Ο κύριος Λίζε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσους ε, μας ε, βοήθησαν στην ε, προετοιμασία αυτού του σχεδίου ψηφίσματος. Νομίζω πως το βασικό μας καθήκον είναι να περάσει αυτό το ψηφίσμα μέσα στι επόμενες εβδομάδες, γιατί όταν είχε συνταχθεί το σχέδιο του ψηφίσματος δεν είχε ληφθεί ακόμα απόφαση από την πλευρά του πρόεδρου Τραμπ και τελικά δεν είναι τόσο δραματικές οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης, τουλάχιστον όπως περιγράφεται από κάποιους, γιατί ε, μία σειρά από πολιτικούς εθνότητες από τις ΗΠΑ είπαν ότι παρόλα αυτά θα παραμείνουν ε, στις δεσμεύσεις τους. Ε, βέβαια, παρόλα αυτά θα πρέπει να υπάρξει μια, πλευρά από τη, μια απάντηση από τη δική μας πλευρά σε σχέση με τα όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ και αυτή η θέση να εκφραστεί στην COP23. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα έγγραφο το οποίο είχε διανύμει ο πρόεδρός μας ε, του, της ομάδας μας, ο κύριος Μάνφρεντ ε, Βέμπερ, όπου ανέφερε το εξής. Τώρα εξαρτάται από την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει ηγετικό ρόλο στην ε, περάσπιση τη συμφωνία του Παρισίου, γιατί είναι μια συμφωνία δίκαια και επειδή διασφαλίζει το μέλλον τόσο του περιβάλλοντό μα όσο και των βιομηχανιών μα. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια του Πρόεδρου τη πολιτική μα ομάδα και θα ήθελα να περιληφθεί και αυτή η αναφορά μέσα στο ε, ψήφισμα. Το ε, πρώτο μας καθήκον είναι να διασώσουμε τη Συμφωνία του Παρισίου, δηλαδή να μην ακολουθήσει κανένας άλλος εταίρος ε, το παράδειγμα του Προέδρου Τραμπ. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ σε καλό δρόμο, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να το αναφέρουμε εμφαντικά, εμφατικά, ότι δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η συμφωνία του Παρισιού. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα όσα συμφωνήθηκαν συμφωνία, να ανταποκρίνονται στους ειδικούς στόχους. Δηλαδή, η ανησυχία μου πια παραμένει. Ε, και σε αυτό βέβαια και στον ανησυχώ ακόμα περισσότερο συνέβαλε και αναφορά του πρώτου Τραμπ. το ότι τα όσα ε, δεσμεύτηκαν να κάνουν συμφωνία του παρουσίου διάφοροι, οι διάφορες χώρες δεν επαρκούν ε, για να επιτύχουμε αυτήν την μείωση κατά δύο βαθμούς ε, Κελσίου. Και δεν ξέρω ούτε καν να φτάνουμε στο 1,5%. Σε κάθε περίπτωση αν αθροίσουμε όλες αυτές τις δεσμεύσεις δεν φτάνουμε στη μείωση κατά 2%. Και βέβαια τα πράγματα έχουν καταστεί ακόμα δυσκολότερα με την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να συγκεντρώσουμε όλους μας του εταίρους ε, για να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η επιπρόσθετη ε, προσπάθεια. Και μέσω του ETS, του Συστήματο Εμπορία Εκπομπών, έχουμε ε, μια δυνατότητα εμείς να αυξήσουμε λίγο το δικό μας στόχο. Και αυτό το στοιχείο, αυτή τη δυνατότητα ενδεχομένω θα μπορούσαμε να την αναφέρουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε με τους εταίρου. Ε, είμαι πάντως φοβισμένος ότι σύντομα θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και ε, ήδη ασκούνται πιέσει. Δηλαδή το 80% όπως ανέφερε και ο ε, Μάνφρεντ Βέμπερ θεωρούν πως η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόβλημα και θα πρέπει να αναλυφθεί δράση για να αντιμετωπιστεί. Οπότε υπάρχει και αυτό, αλλά και δεν γνωρίζουμε και για πόσο πραγματικά καιρό θα παραμείνει πρόεδρο ο κύριο ε, Τραμπ. Δηλαδή δεν θα με εξέπτωει το γεγονό ε, να μην ολοκληρώσει την προεδρική του θητεία. Και αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να ε, κάνουμε τα επόμενα βήματα με του Αμερικανού. Ε, τώρα, για το ΕΛΚ και μετά από τις ε, δηλώσεις που έκανε ο κ. Ε, Τραμπ, το ζήτημα του carbon leakage, ε, της αυτή του, άνθρακα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχει και μια ευκαιρία για τη βιομηχανία, να δημιουργηθούν δηλαδή θέσεις εργασίας που θα είναι και βιώσιμες στο μέλλον. Αλλά υπάρχουν και κάποιες, κάποιοι ε, τομεί, για παράδειγμα όπω τη χαλιβουργία, τη ζωτοποιία ε, ή των λοιπασμάτων που θα αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρί αυτέ τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτούς τους κλάδους μέσω ακριβώς καινοτομιών, μέσω της υποστήριξης έργων τα οποία θα μας επιτρέψουν να παράγουμε τα εν λόγω προϊόντα με μηδενικέ ή εν περιπτώσει σαφώς μειωμένες εκπομπέ ε, άνθρακα. Ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να προέρχεται η σχετική λύση από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να μείνουμε στις διατάξεις προστασίας από το διαρροή άνθρακα, το carbon leakage, γιατί όπως σας είπα υπάρχουν ευκαιρίες οι οποίες ε, δημιουργούνται με ε, αυτή την ανάγκη ε, για τον επιχειρησιακό κλάδο, αλλά από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω υπάρχουν κάποιοι κλάδοι βιομηχανικοί οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να προβούν στις σχετικές μειώσεις. Οπότε αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία με τους συναδέλφους αλλά και με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες και βέβαια και με την Επιτροπή για τη Βιομηχανία, γιατί και εκείνη ασχολείται εντατικά με τον λόγο ζήτημα και αν είναι δυνατό θα πρέπει να λάβουμε πλήρως υπόψη μας τη δική της άποψη έτσι ώστε να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη ε, δυνατή συνένεση το ψήφισμα στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίτερ Για τους σοσιαλιστές εγώ θα πάρω τώρα το λόγο. Ως συν και εγώ του ψηφίσματος αυτού για την COP23. Όπως ήδη υπεθύμησε και η πρόεδρος στην εισαγωγή της, ή και ο Πίτερ Λίζε επίσης, η COP23 στη Βόνη που θα γίνει 6 με 17 Νοεμβρίου υπό την Προεδρία των Ίσων Φίτζη θα λάβει χώρα μέσα σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Γιατί η κόπα αυτή θα λάβει χώρα μετά την απόφαση αυτή του Τραμπ να αποσυρθεί. Και η ανακοίνωση της απόσυρσης αυτής των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων, νομίζω, αν κοιτάξουμε και τις ε, διάφορες αντιδράσεις, ενισχύει τελικά τους υπόλοιπους συνυπογράφοντες και δεν αποδυναμώνει τις υπογραφές τους. Καθ' άλλο. Γιατί από τον Ιούνιο έχουμε διαβάσει ότι πολλοί ηγέτες κατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο το κόσμο επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά τη δέσμευσή τους ώστε να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας ε, του πλανήτη ε, από 2,2 σε 3,6 αν πράγμα το οποίο θα δεν αναλάβουμε τις ε, δικές μας τις ευθύνες, αν δηλαδή δεν τηρήσουμε τόσα λέει η Συμφωνία των Παρισίων. Για να μην υπάρξει λοιπόν αυτή η άνοδο θερμοκρασία, είναι πολύ σημαντικό στο ψήφισμά μα να υπενθυμίσουμε ότι η Συμφωνία των Παρισίων παραμένει ζωντανή Ακόμα κι αν ο Αμερικανικός απομονωτισμός εμφανίζεται, μπορεί να αναδεθεί μια νέα έτσι ηγετική μορφή. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί το νέο ηγέτη που χρειάζεται ο κόσμος για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά κλιματική αλλαγή. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε περισσότερο στο κοινό μας ψήφισμα. Στο κείμενό μας η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει 7 προτεραιότητες για να προχωρήσουν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Πρώτη είναι η δημιουργία καινοτόμων χρηματοδοτικών ε, μέσων για την αντιμετώπιση της κλιματικής ε, αλλαγής. Να υπάρξει ένα νότατόριο ανατόνο άνθρακα και να μεταρρυθμιστεί το σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Δεύτερη προτεραιότητα. Η εγκαθίδρυση μιας πραγματικής κυκλικής οικονομίας και να δοθεί νέα δυναμική στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τρίτη προτεραιότητα. Να σταματήσουν οι επιχορηγήσεις που πηγαίνουν στις ε, συμβατικές ενέργειες, στα ορυκτά καύσιμα δηλαδή, που θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε. Τέταρτη προτεραιότητα περισσότερες προσπάθειες για την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται από τις μεταφορές και τη γεωργία για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020 και το 2030. Πέμπτη προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση να συγκεκριμενοποιηθεί. Πρόκειται για 500 δισεκατομμύρια το χρόνο για τις ανάπτυξη χώρες. Έκτη προτεραιότητα πρόθεση της οικουμενικής πρόσβασης σε ε, βιώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Αφρική, για παράδειγμα, που έχει τεράστιο δυναμικό ανανόσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο όμως δεν εκμεταλλευόμαστε ακόμα. Και η έβδομη προτεραιότητα είναι το πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή την μετανάστευση και πώς θα αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτούς τους μετανάστες λόγω των κλιματικών αλλαγών. Μέχρι το 2050 θα μετακινηθούν 250 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το αγνοούμε πια αυτό. Και το βλέπουμε και σε πολλές αφρικανικές χώρες και της Βόρειας Αφρικής. Πριν από μερικές μέρες ήμουνα στο Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είδα ότι έχουμε όλο και περισσότερους μετανάστες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 40.000 για παράδειγμα από την Νιγερία. Τώρα, μιλάω για αυτές τις μέρες. Μέχρι λοιπόν τις 27 Ιουνίου που έχουμε προθεσμία για να υποβάλουμε τροπολογίες πρέπει να φροντίσουμε να ενισχυθεί το αρχικό αυτό κείμενο. Επιπλέον είμαι ε, συντάκτης γνωμοδότησης για την εφαρμογή της ΚΟΠ στις πόλεις και στην Ήπεθρο και θα ήθελα το ψήφισμά μας ρητά να αναφέρεται στη συνεργασία που πρέπει να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ομόσποδες χώρες, πόλεις και χωριά των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να τηρήσουν τη συμφωνία αυτή που υπέγραψε ο πρόεδρος Ομπάμα. Πρέπει να πούμε στο ψήφισμά μας δηλαδή ότι η Συμφωνία των Παρισίων θα εφαρμοστεί χωρίς τον Τραμπ μεν, αλλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες δε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν φαίνεται ότι έχει βρει με τις 30 Αμερικανικές πολιτείες που είπαν ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία ένα νέο συνομιλητή, παρακάμπτοντας τον Τραμπ. Πρόκειται για μεγάλες πόλεις. <clears throat> Γιατί πολλές από αυτές δεν συμφωνούν με τον Τραμπ. Συνεπώς πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε οι 30 αυτές πολιτείες από τις 50 να, που είναι έτοιμες να μειώσουν κατά 26% τις εκπομπές των ΗΠΑ μέχρι το 2025 να βρεθούν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της COP23 και να είναι πολύ άριθμες εκεί. Αν τα καταφέρουμε θα έχουμε μια πρώτη σημαντική νίκη απέναντι στον ε, Donald Τραμπ. Τώρα, Γκουε. Ο επόμενος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα είναι με τι πολιτική εντολή θα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακόπτη ο Ο συνάδελφο μου που άρχισε, αφήστε τον να ολοκληρώσει. Η κυρία Γκέρλινγκ θα σα συγχωρέσει, γιατί όντω εσεί θα πάρετε το λόγο μετά αντί για τον κύριο Ντάνκαν που δεν είναι εδώ. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριο Χωρίστη. Το θέμα είναι τι πολιτική εντολή θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνοντα στη Βόνη. Το ψήφισμα, κατά τη γνώμη μου, είναι υπερβολικά έτσι δείχνει υπερβολική ικανοποίηση. Τα όμως συμπεριλαμβάνουν οι συμφωνίες που έχουμε μέχρι τώρα δεν φτάνουν για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε οριζόντια όλες αυτές τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με, τη, με το κλίμα. Μόνο έτσι θα έχουμε αξιοπιστία και στις διαπραγματεύσεις μας σε διεθνές επίπεδο, αλλά και απέναντι στους πολίτες. Χρειάζονται αποφασιστικά βήματα στην προσαρμογή, στην βοήθεια για την πραγματική ανάπτυξη, πιο δίκαια ανάπτυξη, να λάβουμε υπόψη μας τις μεταφορές, οδικές, εναέριες και άλλα πράγματα τα οποία ανέφεραν οι συνάδελφοί Πρέπει να πάμε πιο μακριά από την απλή και συνηθισμένη παραδοσιακή ρητορική που κάνουμε σε τέτοιες διασκέψεις. Να μιλήσουμε για την επισητιστική ασφάλεια των αυτοχθόνων πληθυσμών. Και τι κάνει η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας εκπλήξει. Ο πρόεδρος ε, Τραμπ από την αρχή έχει οθετήσει φοβερά πράγματα. Να φτιαχτούν αγωγοί μέσα από γη των αυτόχθονων πληθυσμών ή καταστρέφοντας ε, οικολογικούς χώρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υποστηρίξει πιο αποφασιστικά ένα πρόγραμμα που να είναι και πιο φιλόδοξο. Ευχαριστούμε κύριε Χαρίστη. Τώρα για το ECR η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση ε, που επικράτησε. Όπως ξέρετε, ο κ. Ντάνκρ δεν αλλιώς ε, θα φύγει από το Κοινοβούλιο και γι' αυτό θα είμαι εγώ αρμόδια εκ μέρου του ECR για αυτό το θέμα. Η φιλοδοξία σε αυτό το σχέδιο του ψηφίσματο είναι πολύ καλή. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω την πρόκληση που υπάρχει. Αυτό θα πρέπει να είναι συνδυτό στο Κοινοβούλιο. Είναι σωστό να υπάρχει ιεράρχηση ε, να υπογραμμίζεται η ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχουν ε, διατομεακές ε, ε, παρεμβάσεις, να αναπτυχθεί η διπλωματία, κυρίως λόγω της απόφασης του Πρόεδρου Τραμπ. Επίσης, χαιρετίζω αυτό που ελέγχθη σχετικά με τον, τη διεθνή αεροπλοεία. Πάρα πολλοί εργάζονται πάνω σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπας περιπτώσει, έχω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την σύνταξη του κειμένου. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα εκπομπών που πρέπει να επισημάνουμε. Παρότι λοιπόν το 2018 ο διάλογος μας προσφέρει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε τότε την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί σε σχέση με την πρόοδο για τους στόχους ε, που έχουν καθοριστεί. Εγώ παρόλα αυτά λέω ότι θα πρέπει να προσέξουμε την παράγραφο 7 που αφορά ε, τους στόχους του 2020. Εκεί γίνεται λόγος ε, για επενδυτικούς κύκλους. Για μένα η για την επόμενη συνδιάσκεψη είναι διαφάνεια, ευκρίνεια, να κατανοήσουμε τους στόχους έτσι ώστε να μπορούμε και να αξιολογήσουμε τις ε, καταβαλλόμενες προσπάθειες. Αν δεν γίνει αυτό, τότε ε, δεν θα μπορέσουμε και να προχωρήσουμε. Επίσης, ε, αυτό που λέγεται για τη διαφοροποίηση των ρηκτών καυσίμων, παραγράφος 13, εκεί θα ήθελα να υπάρχει κάποια αναφορά στα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων και αυτά θα πρέπει να είναι συμβατά με τους υπάρχοντες ορισμούς. Και αναφέρω επίσης ότι θα πρέπει να γίνεται και λόγος για την ανεπάρκεια. Αυτό αναφέρεται στις δεσμεύσεις του G20. Υπάρχει δέσμευση ενός μηχανισμού για την ενίσχυση περίπου γίνεται λόγος για 100 100 δισεκατομμύρια. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί πρόβλημα. Η σημαντική μείωση στην συνεισφορά των ΗΠΑ καθιστά απαραίτητο για την Ευρώπη να αυξήσει τη συνεισφορά τη προ το Ταμείο του Πράσινου Κλίματος. Η αποφάσεις ε, σχετικά με την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σίγουρα παίζουν ρόλο. Δεν στηρίζω αυτό που λέγεται για το ότι θα πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετη υποστήριξη. Δεν υπάρχει σαφής ορισμός για το τι πρέπει να περιλαμβάνεται. Ε, όσον αφορά όμως τις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές λένε ότι η βοήθεια θα πρέπει να δίνεται και σε συνδυασμό με τους ε, στόχους για την ανάπτυξη. με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις ε, της ΚΟΠ ε, θεωρώ ότι το κείμενο θα πρέπει να τροποποιηθεί. Αυτό προτείνεται. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να εισαχθεί ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, οι φόροι αυτοί συμφωνούμε επί της αρχής, αλλά ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να ισχύει σε παγκόσμια κλίμακα. Και όσον αφορά άλλα θέματα, ε, θα καταθέσω τροπολογίες ε, σχετικά με το Brexit και επίσης ε, θα θελήσουμε να υπογραμμίσουμε και τη συνέχεια της συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις κλιματικές παρεμβάσεις. Κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν πολλές δεσμεύσεις ουσιαστικές πέμπτος ε, προϋπολογισμός ε, για τον Ανθρακά καθορίζει συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2030. Και τέλος, ε, κάποια λόγια θα ήθελα να σας πω για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χωρίς να υπάρχει ισορρευτική δέσμευση, οι Ηνωμένε Πολιτείε σίγουρα υπονομεύουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι μέχρι το 2050. Αλλά επίσης όλα αυτά είναι επιζήμια και βραχυπρόθεσμα γιατί η αξιοπιστία των Παρισίων είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει η υποστήριξη των ΗΠΑ, νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τη σωστή προσαρμογή που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το δυναμισμό που στριλατήθηκε στο Παρίσι. Αφήσουμε τον φόρο των χρηματοψηφιωτικών συναλλαγών. Θέλουμε πρακτικέ λύσει για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση σε σχέση με το υπάρχον ταμείο και αυτό θα πρέπει να γίνει και αρκετά γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γκέρλινγκ. Από το Άλντε κανείς. Ο Μάρκο Αφρόντο τώρα, εκ μέρους των Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγα θα πω γιατί η έκθεση μοιάζει να είναι ολοκληρωμένη και ίσως ε, να μην ε, δείχνει το ότι επήγει το όλο θέμα. Ε, η έκθεση Όσον αφορά την έκθεση νομίζω ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο για να επιτύχουμε του στόχου του Παρισιού. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να επιτύχουμε το στόχο τη μείωση του 2%, πόσο μάλλον του 1,5%. Θα ήθελα λοιπόν να πω κάποια λόγια ε, που αφορούν όχι μόνο στο ότι πρέπει να δράσουμε, αλλά και στο ότι πρέπει να βιαστούμε. Κάτι συγκεκριμένα που αφορά στο σημείο υπαριθμών 6, όπου για μία ακόμη φορά χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το όλο θέμα γίνεται ένα βήμα προς τα εμπρός ε, και ε, στη Συμφωνία του Παρισιού αναφέρεται ο στόχος ε, να επιτευχθεί η ισορροπία όσον αφορά στις ανθρωπογενείς εκπομπές και στην απορρόφηση των εκπομπών από απορρόφηση των εκπομπών από συλλέκτες αερίων του θερμοκηπίου. το να βασιζόμαστε μόνο σε αυτό για να επιτύχουμε τους στόχους μας, αυτό είναι κάτι που σημαίνει ότι απλά αναβάλουμε την όλη κατάσταση ε, και αυτό θα έχει αρκετά σοβαρές συνέπειες, ενώ πρέπει να δουλέψουμε πολύ πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, η ε, Συμφωνία των Παρισιού, του Παρισιού ε, δεν αναφέρει τόσο συχνά το θέμα της οικονομίας χαμηλού άνθρακα, που είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Όσον αφορά το θέμα των ΗΠΑ, της τελευταίες ημέρες υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω με ικανοποίηση ότι αυτά όλα δεν δημιούργησαν μόνο ε, μία χιονοστιβάδα, αλλά ε, κατ' ουσίαν και δυνάμωσαν εκείνους ε, τη θέληση εκείνων που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Παρισιού. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Κίνα αν θέλουμε να καλύψουμε τη θέση που αφήνουν κενή οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Και θα ήθελα και να προσθέσω ότι ε, στη Συμφωνία του Παρισιού γίνεται μόνο ε, μία αναφορά στο μηχανισμό loss and damage και αναφέρεται εκεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ο μηχανισμός αλλά θα συζητήσουμε αργότερα. Στην COP22 δεν συζητήθηκε το θέμα. Από ό,τι φαίνεται ούτε και στην COP23 αναφέρεται ως προτεραιότητα. Είναι όμως ένα σημαντικός μηχανισμός γιατί μιλάμε για χώρες ε, του ειρηνικού που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, υφίστανται όλες αυτές τις συνέπειες. Είναι ένας οικονομικός ε, μηχανισμός που θα πρέπει να εγγυάται το τι είναι εφικτό. Βεβαίως ε, είναι ένα θέμα το οποίο, όπως σας λέω, δεν μπορούμε να το αφήσουμε με μια απλή αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το εξετάσουμε σε βάσος και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε το θέμα αυτό να το εξετάσουμε στην COP23 στη Βόνη. Ευχαριστούμε κύριε Φρόντε. Ο κύριος Πεντιτσίνη τώρα, εκ μέρους του Διευθυντή. Πρόεδρε, ζητήσαμε από την Επιτροπή να μας πει τι σκοπεύει να κάνει για να εγγυηθεί ότι η συνδιάσκεψη της Βόνης θα σημειώσει ουσιαστική πρόοδο σε σχέση με τη Συμφωνία του Παρισιού. Ε, και ζητήσαμε να γνωρίζουμε και πώς θα μετρηθεί η πρόοδος. Επίσης, ε, κατά πόσον θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, ε, γιατί ο στόχος είναι 100 δις το χρόνο μέχρι το 2020. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, πολύ πιο σημαντικό, μια ερώτηση που γίνεται όχι τόσο στην Κομισιόν, αλλά στα κράτη-μέλη πρέπει να διερωτηθούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί η σημαντική πρόοδος. Και εμεί λοιπόν συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να προσθεθεί κάτι που να αφορά στι ΗΠΑ. Δεν θέλουμε όμω μετά την παρέτηση των ΗΠΑ και την αποχώρησή του από την ε, Συμφωνία του Παρισιού, οι ΗΠΑ να γίνουν ο αποδιοπομπαίο τράγο και όλοι να κρυφτούν πίσω από αυτό αυτόν τον τράγο ή από τον κύριο Τραμπ. Είναι πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, εκείνο που ισχύει είναι ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λόγια τα πάνε πάρα πολύ καλά, λένε πολλά υπέρ της κλιματικής αλλαγής, αλλά στην πράξη, κατ' ουσίαν, ε, εξακολουθούν να προάγουν την έρευνα που έχει σχέση με το πετρέλαιο. Άρα δηλαδή ε, ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά. Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία ε, υπερισχύουν ε, των λέξεων και των φράσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλοί κρύβονται πίσω από τον Τραμπ αντί να λάβουν μόνοι τους τις ευθύνες τους. Και εσείς ε, κύριε Πρόεδρε είπατε προηγουμένως ότι η δική σας ομάδα συμφωνεί ε, να ε, εξαλειφθούν οι χρηματοδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα αλλά στη δική μας την ομάδα υπάρχουν εκπρόσωποι κυβερνήσεων οι οποίοι κατά περίεργο τρόπο λένε τα ίδια που λέτε κι εσείς αλλά επί της ουσίας κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Η Ιταλία, παραδείγματο χάρη, επένδυσε 80 εκατομμύρια ευρώ στο Green Fund, στο Πράσινο Ταμείο, αλλά παράλληλα 14 δις ευρώ τα δαπανά για να στηρίξει τα ορυκτά καύσιμα. Νομίζω ότι θα πρέπει πότε να δούμε τους ε, σκελετούς που έχουμε στην ευρωπαϊκή ντουλάπα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μιρέη έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της ανθρωπότητας σήμερα. Παρ' όλα αυτά, λυπάμαι πολύ που μιλάμε τόσο πολύ για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συμφωνία. Με η Συμφωνία αυτή μιλάει για συγκεκριμένες δράσεις σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να βρούμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης ε, στη δράση για το κλίμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είπαν ότι θέλουν να αποχωρήσουν από τη Συμφωνία των Παρισιών. Παρόλα αυτά συμμετέχουν στη σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή ή ακόμα και στον ΙΚΑΟ ή στον, ε, Ευρωπαϊκό, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Άρα εδώ δεν πρέπει να πιέζουμε τις αρμοδιότητες των χωρών. Με το ψήφισμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την απογοήτευσή του απέναντι στον ΙΚΑΟ, στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και το ίδιο κάνει και για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δίνει την προτεραιότητα στην κλιματική διπλωματία αυτό όμως σημαίνει ότι πλήττεται τη δυνατότητα των χωρών μελών και τις δικιάς τους δράσεις στα πλαίσια αυτών των διεθνών οργανισμών, γιατί θεωρείται ότι παρεμβαίνουν και ότι δεν θα έπρεπε. Οπότε στις υπανάπτυξη χώρες ε, κυρίως θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρώτα απ' όλα. Η δικιά μου χώρα, η Γαλλία, ήδη είναι καθαρός εισφορέας με πολλά δισεκατομμύρια υπέρ της δράσης για το κλίμα. Τέτοιες επενδύσεις δεν είναι δυνατόν να γίνονται χωρίς τακτικό και αυστηρό έλεγχο. Αλλιώς χάνουμε την αξιοπιστία μας. Ευχαριστούμε. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Έχω εδώ τον κύριο Μπάξο νομίζω. Έτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω αρχικά ότι συμφωνώ Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισίου. Ωστόσο, ε, δεν συμφωνώ με το να αντιμετωπίσουμε ως ε, κάτι το δευτερεύον ε, την απόσυρση ουσιαστικά την αποχώρηση από τη Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο δεύτερος ε, μεγαλύτερος ρηπαίνων παγκοσμίω και αυτό έχει και επιπτώσει σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. του στόχου δηλαδή ε, της ε, μείωσης σε σχέση με τα βιομηχανικά επίπεδα της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι δυσκολότερο λοιπόν να επιτύχουμε αυτό το στόχο. και πριν από τη Συμφωνία του Παρισιού είχε θεωρηθεί ότι πράγματι είναι καλό να είμαστε φιλόδοξοι και θα πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο όμως ε, κάποιοι είχαν αναφέρει επίσης ότι θα επιτύχουμε τους ε, στόχους μας εφόσον και μόνο εφόσον οι ε, κύριοι ρηπαίνοντε αναλάβουν νομικά δεσμευτικέ υποχρεώσει. Τώρα λοιπόν ε, Θεωρούμε πως υπάρχει μια ιστορική συγκυρία γιατί ε, ακριβώς υπάρχουν τέτοιου είδους νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις ε, και εγώ είχα ρωτήσει και τον Επίτροπο ε, Γανιέτε πώς θα μπορούσαν να να ανταποκριθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, στι υποχρεώσει που είχε αναλάβει ο πρόεδρο ε, Ομπάμα στο ενδεχόμενο προεδρία του πρόεδρου Τάμπ, γιατί ήμουν ένα από του λίγου που θεωρούσε ότι υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο. Άρα λοιπόν, μου είχε πει ότι οι εν λόγω υποχρεώσει παραμένουν νομικά δεσμευτικέ για όλα τα κράτη που συμμετέχουν, τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, τελικά είδαμε στο Παρίσι ότι δεν είναι νομικά ή λόγω υποχρεώσεις. Από εκεί και μετά θα ήθελα να θέξω δύο σημεία. Έως ε, τις 27 ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ε, βάλουμε ε, τροπολογίες. Οπότε εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια αναφορά στις ΗΠΑ. Στο σημείο 4 βέβαια αναφέρεται ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνένεση σε ό,τι αφορά την επίτευξη των σχετικών στόχων, ε, γεγονό το οποίο επιχαίρουμε, παρά των πολιτικών μεταβολών ε, που έχουν λάβει χώρα. Ότι δηλαδή παρά αυτέ τι μεταβολέ, ε, τα διάφορα συμβαλωμένα μέρη, διάφορε χώρε μένουν στι υποχρεώσει του. Εντάξει, επειδή ω τι 27 θα έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε τροπολογίε, εγώ θα ήθελα ε, να, ε, ε, το συγκεκριμένο σημείο να ενημερωθεί, να επικαιροποιηθεί ουσιαστικά, δηλαδή να κάνουμε μια συγκεκριμένη αναφορά ότι τουλάχιστον προσωρινά οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποχωρήσει από τη συμφωνία και κατά συνέπεια θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι ρεαλιστικά επιτεύξιμη η σχετική στόχη. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Η κυρία Παρμπραμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλησπέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, ούτω ώστε να ανταλλάξουμε απόψει μετά από τις τελευταίε εξελίξεις συμπεριλαμβανμένες της ανακοίνωσης της κυβέρνηση Τράπο, ότι δηλαδή προτίθεται να αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισίου. Ε, πρόκειται μόνο για μια δήλωση πρόθεση από την πλευρά των ΗΠΑ. Δηλαδή προ το παρόν παραμένει συμβαλλόμενο μέρο ε, και τη ε, σύμβαση και τη Συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το σχέδιο ψηφίσματο το οποίο προτείνει το Κοινοβούλιο, θεωρούμε πως είναι ε, πραγματικά μια πολύ ε, ισορροπημένη ε, και διεξοδική αναφορά των προτεραιοτήτων. δηλαδή, περιλαμβάνει ζητήματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε στο πλαίσιο της COP23, αλλά και ζητήματα που θίγουν περαιτέρω χώρες. ζητήματα τα οποία θα είναι εξαιρετικά σημαντικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των όσων συμφωνήθηκαν στο Παρίσι. Αυτό που βλέπουμε ως δηλαδή αντιδράσεις ανά τον κόσμο ε, απέναντι στην ε, ε, απόφαση της κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι δεν υπήρξε αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση την οποία φοβόμασταν. Δηλαδή ότι κάποιες χώρες θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της κυβέρνησης Τραμπ. Αντιθέτως, ενισχύθηκε η αποφασιστικότητά τους να ε, ε, μείνουν στις ε, δεσμεύσεις τους. Και μάλιστα υπάρχουν πολλοί φορές τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή πολιτείες των, Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρήσεις και άλλοι φορεί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους σε αυτούς τους στόχους και δήλωσαν ότι δηλαδή θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές τις εθνικές συνεισφορές που είχαν καθοριστεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, και την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ε, και για μία ακόμα φορά ε, πόσο διατεθειμένο είναι και το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιτύχουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του 40% έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο σχετικό στόχο. Ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα αυτός ο στόχος, γιατί συμφωνώ με όσους είπαν ότι η διευκόλυνση του διαλόγου για τον χρόνο θα αποτελέσει και μια ευκαιρία προκειμένου να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει σε ό,τι αφορά την επίτευξη των σχετικών στόχων. Ποιοι είναι δηλαδή οι μηχανισμοί που έχουμε δημιουργήσει για την επίτευξη των στόχων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους στόχους ε, για τις COP23. Ε, Σίγουρα δεν θα είναι ορόσημα, αν θέλετε, ή κάποια υπέρβαση αυτή η COP23. Ε, εκείνο που θέλουμε να επιτύχουμε μια σταθερή πρόοδο σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, ή το χάρτη πορείας που είχε καθοριστεί στη Συμφωνία του Παρισίου. Και θα πρέπει ενδεχομένω να συγκεκριμενοποιήσουμε και τις προσδοκίες που έχουμε. Δηλαδή δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει ακριβώς το τι θα πρέπει να γίνει. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι ε, να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο μετριασμό, αυτό το mitigation και από εκεί και μετά τα ζητήματα αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα μεταφορά τεχνολογία και τεχνογνωσίας, δημιουργία ικανοτήτων και ούτω καθεξής. Με αυτή λοιπόν τη διευκόλυνση του διαλόγου θα διασφαλίσουμε τον παγκόσμιο χαρακτήρα τη δέσμευση. Πέραν αυτών των στόχων τη COP23 θα πρέπει να εργαστούμε και στον χώρο non-state space δηλαδή στο ε, πλαίσιο τη ε, ατζέντα του θεματολογίου για την παγκόσμια δράση. Έχει, έχει λάβει τώρα υψηλότερη σημασία γιατί για να επιτύχουμε εδώ του στόχου ε, και το όρομα τη Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να υπάρξει κοινή συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών. Το εγώ ε, θα ήθελα να υπάρξει μια επικυρωποίηση του σχεδίου ψηφίσματος ε, ε, προκειμένου να αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτή την απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ. Και όπω γνωρίζετε το Συμβούλιο τη Δευτέρα υιοθέτησε συμπεράσματα όπου ακριβώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για αυτή την απόφαση τη κυβέρνηση Τραμπ και επανέλαβε την πρόθεσή του να ανταποκριθεί στις εθνικές συνεισφορές ή τις συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλάβει, αλλά και προκειμένου να αναβαθμίσει τη συνεργασία και να επιτείνει τη συνεργασία του με του ε, διεθνεί εταίρου, ούτω ώστε ε, να επιτευχθούν περισσότερα στο πλαίσιο τη ε, κλιματική διπλωματία. Και εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή ακριβώ αυτό θα να κάνουμε. Δηλαδή, ο δικό μα Επίτροπο αποφάσισε με τον Υπουργό του Καναδά και τη Κίνα, του αρμοδίου, να υπάρξει μια κοινή συνάντηση στην ΤΑΒΑ ε, Ενδεχομένω ε, ε, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών φέτος, προκειμένου ακριβώς να ενισχυθεί η Συμφωνία, η Παγκόσμια Συμφωνία σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας, όχι μόνο με τις μέγιστες οικονομίες, δηλαδή του G20, αλλά της ΑΚΕ, της Αφρικανικής Ένωσης και άλλους. Άρα λοιπόν θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχίσει αυτή η η όθηση που έχει δοθεί ε, και προκειμένου όλοι οι εταιρείε να ανταποκριθούν στα όσα συμφωνήσαμε. Ε, και νομίζω πως είναι ε, χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν ισούται με όλους τους εταίρους μας από τις ΗΠΑ. Υπάρχει για παράδειγμα ο κυβερνήτης Μπράουν της Καλιφόρνια, ο οποίος θα είναι ο κοδεσπότης αν της ε, συνέλευσης της ε, Παγκόσμιας Συνεδρίας για κλιματική αλλαγή του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τόσα μας είπατε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξαναβρεθούμε βέβαια ακριβώς στη Βόνη για αυτήν την COP23. Προς ενημέρωσή σας, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξή υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 27 Ιουνίου στις 11 εξέταση των τροπολογιών στις 30 Αυγούστου 2017, ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΝΒΗ 7 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Προτείνω να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τώρα, που είναι ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την σχέση του και τη σύνδεση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αντίστοιχο της Ελβετίας. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Η κυρία Γκράτς. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή για μια ανταλλαγή απόψεων για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για να κάνουμε απολογισμό του τι συμβαίνει και υπάρχουν οι τελευταίες εξελίξεις ε, που αφορούν γενικότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Πώς ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι το σύστημα αυτό της ανταλλαγής των δικαιωμάτων εκπομπών, το ETS, είναι το πιο αποτελεσματικό για να περιστούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Τώρα λοιπόν δουλεύουμε πάνω στην επόμενη αναθεώρηση αυτού του συστήματος για να είμαστε σωστά εξοπλισμένοι το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει λοιπόν την εμπειρία αυτού του συστήματος ε, και μέχρι τώρα είναι ο χώρος όπου χρησιμοποιείται ευρέως αυτό το σύστημα. Αλλά πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης να στηρίξει την εφαρμογή ε, μιας εύρυθμα λειτουργούσα αγοράς άνθρακα και αυτό μέσα από το σχεδιασμό του συστήματος ETS σε τρίτες χώρες με στόχο βεβαίως να υπάρχει κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, μια μεγαλύτερη αγορά άνθρακα, έτσι ώστε να υπάρχουν και ίσοι όρια ανταγωνισμού. Αυτή είναι η μακροχρόνια στόχοι πολιτικής που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που σε μεγάλο βαθμό τους στόχους αυτούς τους συμμερίζεται η διεθνής κοινότητα, διότι θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να επιδιωχθούν οι στόχοι του Παρισιού. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, εμείς καθορίσαμε μία βάση για να συνδέσουμε ένα συγκεκριμένο άρθρο, το υπαρτμόν 25 της οδηγίας ETS, που προσφέρει τη δυνατότητα το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδυαστεί με άλλα συστήματα ανταλλαγής εκπομπών, δικαιωμάτων εκπομπών, υπό την προπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν και συγκρίσιμα συστήματα. Να σας υπενθυμίσω ότι το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει και για την ε, ε, Νορβηγία, το Λίχτενστάιν, την Ιρλανδία. Βεβαίως η Ελβετία είναι η μόνη χώρα ε, όπου δεν ισχύει το σύστημα ETS και η Ελβετία έχει το δικό της το σύστημα το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται το 2008. Εάν λοιπόν συγκρίνουμε με την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συγκρίνουμε το ελβετικό σύστημα, έτσι κι αλλιώς η ελβετική αγορά είναι πολύ πιο μικρή. Έχει το δικό της το ενεργειακό μείγμα που βασίζεται σε υδρογόνο και σε πυρηνική ενέργεια. 5 εκατομμύρια τόνοι σε σχέση με τα 2 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πέρα από την τάξη μεγέθους, αν δει κανεί τα βασικά χαρακτηριστικά του ελβετικού συστήματος, αυτά μοιάζουν πολύ με τα χαρακτηριστικά που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ε, δεσμευτική η εφαρμογή αυτού του συστήματος στον βιομηχανικό τομέα. Υπάρχει παρεμφερής ρόλο στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και πάρα πολλά. Υπάρχουν βέβαια και διαφορές, ε, αλλά θα επανέλθω σε αυτό, αφορά την αεροπλοεία. Και ακριβώς αυτό κάναμε εμείς όταν εξετάσαμε τη Συμφωνία Σύνδεσης. Για όλους αυτούς τους λόγους η Ελβετία ήταν υποψήφια στο να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σύνδεσης των συστημάτων, εκτός το ότι μιλάμε και για μια ευρωπαϊκή χώρα με την οποία έχουμε πολύ στενούς οικονομικούς δυσμούς, προφανώς και αυτό έπαιξε ρόλο για να ληφθούν υπόψη στο κατά πόσον θα συνδεθούν τα συστήματα, έχοντας αυτά κατά μετά από πρόταση της Κομισιόν, το Συμβούλιο τον Δεκέμβρη του 2010 ενέκρινε μία απόφαση που έδινε, εξουσιοδοτούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Σουηδία. Και ακριβώς αυτό συνέβη πριν από κάποια χρόνια. Και αυτό πάλι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων και διαπραγματεύσεων με την Ελβετία. Όπως είπα προηγουμένως, η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει είναι στην αεροπλοεία. Εκεί η αεροπλοεία προφανώς είναι σε μεγάλος συνεισφέρον στο ε, φαινόμενο του θερμοκηπίου στη χώρα. Εμείς ε, θελήσαμε να υπάρχει ένα προαπαιτούμενο που να αφορά στην αεροπλοεία για να συνδεθούν τα δύο συστήματα ETS. Και τελικά αυτό έγινε αποδεκτό. Η Ελβετία δέχτηκε να ε, Ευχαριστώ δώσει δική μέρημνα στην αεροπλοεία και λόγω της πολιτικής ε, συμφωνίας που επιτέχθηκε ήδη ε, λειτουργεί το όλο θέμα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό επίτευγμα. Όπως και το Ευρωπαϊκό ΙΤΕΣ και το Ελβετικό αυτή τη στιγμή αναθεωρείται ε, για το 2013 και μετά οι αλλαχές που προβλέπονται, αυτές οι αλλαγές θα τις δούμε πιο προσεκτικά, έχουν στόχο να διασφαλίσουν την την συμβατότητα με το δικό μας, με το ε, ETS ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όμως ε, και ένας μηχανισμός αναθεώρησης που θα μπορεί κανείς να αναθεωρήσει το σύστημα από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί και το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της, επί της ουσίας τώρα. Όπως βλέπουμε από την ίδια την συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις έγιναν ε, με βάση ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των δύο συστημάτων και βασικά κριτήρια, βασικές αρχές, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές ε, να μπορούν και οι δύο να είναι πεπισμένες για τη συγκρισιμότητα των συστημάτων. Αυτό το βλέπετε στο παράρτημα. Υπάρχει πράγματι η συγκρισιμότητα και όπως ανέφερα και προηγουμένως η ιδέα είναι να υπάρχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα αναθεωρήσεις των συστημάτων. Οι διαπραγματεύσει ε, ε, ολοκληρώθηκαν στο 2015 και στο πλαίσιο του COP21. Τότε ξεκίνησε και ο σχεδιασμός μιας συμφωνίας για να τεθεί σε ισχύ το 2016. οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τότε, όπως σας είπα, γιατί αποτελούν ένα κομμάτι του ευρύτερου πακέτου των διαπραγματεύσεων με την Ελβετία. Ε, όπως ξέρετε, κάποια στιγμή υπήρξε μια αναστολή των πάντων και γι' αυτό ίσχυσε η αναστολή και για το ETS μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελβετία. Έγινε νέα πολιτική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποια στιγμή αποφασίστηκε αυτό το σύστημα να αποσυνδεθεί από το υπόλοιπο πακέτο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε να προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα και αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή υπάρχει μια πρόταση ε, για να ληφθεί μια απόφαση για υπογραφή και για να εξαρθούν και, και για να ολοκληρωθεί και όλη η συμφωνία. Η απόφαση για την ολοκλήρωση θα επιτρέψει να κατατεθεί όλο αυτό για κύρωση και μετά η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή από τη στιγμή που η συμφωνία έχει πάει στο Συμβούλιο και εφόσον έχει υπάρξει και η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτή τη φάση, θα ήθελα να σας πω ότι θα κριθεί απαραίτητο να υπάρξει και τεχνική εργασία, έτσι ώστε και οι δύο πλευρές ε, να είναι έτοιμες για τη σύνδεση των συστημάτων. Ε, να γίνει δουλειά όσον αφορά ε, τα μητρώα, αυτή είναι πολύ σημαντική δουλειά και όπως σας είπα και προηγουμένως, επειδή υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη ότι το σύστημα ETS στην Ελβετία θα καλύπτει και την αεροπλοεία. Αυτό είναι σημαντικό με την αεροπλοεία. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η πρώτη συμφωνία σύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό ETS και ένα άλλο ETS. Είναι λοιπόν ορόσημο αυτή η συμφωνία και είναι και μοναδική θα έλεγα γιατί το ελβετικό ETS και αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι μοναδικό. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο, μήνυμα δραστηριοποίησης αλλά και πολιτικής δέσμευσης εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχοντας κατά αυτά που ελέγχθησαν προηγουμένως, ε, αυτό το μήνυμα είναι πολύ σημαντικό και για ευρύτερα, για ολόκληρο τον κόσμο, σε διεθνή κλίμακα. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λορόνς Γκράς. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντάλη τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ την κυρία Γκράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Θέλω όμω τώρα να αναφερθώ στο τελευταίο που είπε. Εγώ νομίζω ότι η σύνθεση αυτή με την Ελβετία είναι ένα σημαντικό βήμα ένα πρώτο σύνδεσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων με την έξω αγορά. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Μήπως η σύνδεση αυτή γίνει και με άλλες περιπτώσεις. Όχι μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης. Πολλά είναι τα ωφέλη κατά τη γνώμη μου. Είδα τη σύνδεση του συστήματος αυτού με το ελβετικό σαν μια ευκαιρία και σταθερότητα. Κάτι το οποίο θα βελτιώσει την βεβαιότητα για τους επενδυτές, οι οποίοι θα ξέρουν ότι έχουν ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζεται από μια μεγαλύτερη αγορά. Το βήμα αυτό το βλέπω όπως σας είπα ως το πρώτο προς μια διεθνή συνεργασία και ως δέσμευση σε μια μακροχρόνια περιβαλλοντική πολιτική που θα μας βάλει στην πρώτη γραμμή παγκοσμίω. Φυσικά υπάρχουν και κίνδυνοι από κάτι τέτοιο. Και θέλω να καταλάβω κάπως καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι βήματα περιλαμβάνονται, τι βήματα έχουν αναλυθεί για να αντιμετωπιστούν τέτοιες ανησυχίες. Δύο κυρίως. Πρώτον, ότι η σύνδεση αυτή μπορεί να επηρεάσει την ε, διανομή και την κατανομή και ότι μπορεί να επηρεαστούν οι τιμές. Και το άλλο θέμα είναι η αστάθεια του συστήματος στις τιμές από το άλλο σύστημα ακριβώ. Και τι μέτρα λαμβάνοντας τη σύνδεση αυτή δεν θα υπονομεύσει περιβαλλοντικές ε, πολιτικές όσον αφορά την τιμή άνθρακα. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή τι αντισταθμιστικά μέτρα λαμβάνονται ώστε το σύστημα να λειτουργήσει καλά, χωρίς προβλήματα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λενόνσκας, παρακαλώ. Για να απαντήσει, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για την στήριξή σας που συμφωνείτε για την αρχή αυτή της σύνδεσης και το ότι αυτό μας βάζει στην πρώτη γραμμή. Είναι κάτι που και εμείς το έχουμε υπόψη μας. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω και κάτι, γιατί τα θέματα που πολύ σωστά υπογραμμίζετε ως δεχόμενους κινδύνους ισχύουν πράγματι γενικά όταν μιλάμε για τέτοια σύνδεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι ελάχιστη εξαιτία του μεγέθους της αγοράς, της ελβετικής αγοράς και τις διαφορές που υπάρχουν στις τιμές. Έχοντας αυτό υπόψη λοιπόν δεν βλέπουμε πραγματικά αν ελοχεύει κίνδυνος, μάλλον καθόλου. Και βέβαια υπάρχουν μηχανισμοί στο σύστημα που μας επιτρέπουν να αναλάβουμε δράση αν δούμε να επαληθεύεται κάποιος κίνδυνος. Αρκετά πίθανο κατά τη γνώμη μας. Η συμφωνία, ας πούμε, αναφέρει διάφορες δυνατότητες διακοπής ή και παύσης της συμφωνίας σε κάποιες περιπτώσεις. Για την αστάθεια στις τιμές τώρα και τη διανομή δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή τη συγκεκριμένη αγορά τουλάχιστον την ελβετική. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άλλους κανείς? Όχι? Ωραία. Τότε περνάμε στο επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Και αυτή είναι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, γιατί στις περιόδους 2008-2011 και 2011-2014. Θα δώσω συνεπώς το λόγο στον κύριο Λέγκεντοφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει το θέμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you uh, very much, and thanks for uh, the opportunity. Σας ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτήν την έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής. Αφορά δηλαδή την μεταφορά στην εθνική νομοθεσία αλλά και την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας για την περίοδο 2008-2014, δηλαδή μια εξαετή περίοδο. Και όπως σας είπα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της ε, οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, αλλά και την εφαρμόγη των διατάξεων ε, επιτόπου δηλαδή από τα κράτη-μέλη. Αξιοποιήσαμε μία σειρά από πηγές ε, προκειμένου να συνθέσουμε αυτή την έκθεση, δηλαδή βασιστήκαμε στα δεδομένα των κρατών που μας παρέχαν στο πλαίσιο ενός κραταμένου ερωτηματολογίου, αλλά και περαιτέρω πηγέ. Ε, ειδικότερα, για παράδειγμα, το fitness test το οποίο είχαμε ε, εξάγει το 2014, το fitness tech, ε, σε σχέση και με αυτή και με μια άλλη οδηγία, σε σχέση δηλαδή ακριβώς με την αποτελεσματικότητα αλλά και την προστιθέμενη αξία των διατάξεων της παρούσας και ε, περαιτέρω οδηγιών. Βασιστήκαμε λοιπόν στα στοιχεία και ε, αυτής της ε, fitness tech. τώρα, ε, ποιος ήταν ο βασικός στόχος η, αυτής της η πρόληψη της συμπερίληψης επικίνδυνων αποβλήτων και γενικά αποβλήτων ε, στην κατασκευή των αυτοκινήτων. Ε, πρόκειται για την προώθηση ανακυκλωμένων υλικών στα οχήματα και ε, την κατάλληλη ανακύκλωση των υλικών του ειδικότερα όταν αυτά αποσύρονται από την κυκλοφορία. Ε, και προκειμένου να γίνεται δηλαδή η συλλογή των πολύτιμων υλικών τους ε, σε εγκεκριμένα σημεία ή συγκεκριμένε εγκαταστάσει ανακύκλωση. Ακριβώ προκειμένου τα εν λόγω υλικά να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται ή και σε ορισμένε περιπτώσει να λαμβάνονται αυτούσια από αυτά τα οχήματα. Ε, και αναφέρουμε συγκεκριμένα ότι στόχη είναι το 95% των οχημάτων, ε, των οικοτών οχημάτων να ανακυκλώνονται και το 85% να ανακυκλώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται. Εδώ έχουμε να κάνουμε με οδηγίες ε, που είχαν ε, ξεκινήσει, ε, η οδηγία που ξεκίνησε την εφαρμογή το 2000, υπήρχαν κάποιες διαδικασίες κατά παράβαση, κατά κρατομελών που δεν είχαν μεταφέρει σωστά τις διατάξεις στην εθνική νομοθεσία. Αλλά επιλύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Χρειάστηκε βέβαια σε μια στην άλλη περίπτωση να το σφίγμα και ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουν επιληθεί τα προβλήματα της μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ...επί τόπου πραγματική εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας στα κράτη-μέλη. Η έκθεση καταδεικνύει ότι υπήρξε μια γενικά καλή εφαρμογή, ότι δηλαδή υπάρχουν καλές πρακτικές που ε, χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη, δηλαδή ένα πολύ πυκνό δίκτυο επεξεργασίας, δηλαδή με 13.000 εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ε, για αυτά τα οχήματα. Υπάρχουν και καινοτόμες τεχνολογίες, ε, για τη διασφάλιση ακριβώς ε, τα υψηλά ποσοστά επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και όπως αναφέρουμε και στο τέλος της έκθεσης υπάρχουν μία σειρά από προκλήσεις που κρεμούν ακόμα, ε, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι ένα σημαντικό αριθμό οχημάτων που φτάνουν στο, κύκλο, στο τέλο του κύκλου ζωή του που δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Δηλαδή τα οποία ε, δεν βρίσκονται πλέον σε κυκλοφορία, δεν είναι πλέον ε, ταξινομημένα με βάση την πινακίδα τη κυκλοφορία, αλλά δεν έχουν ταυτόχρονα φτάσει σε μία εγκατάσταση. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν έχει γίνει κάποια ε, παράνομη εξαγωγή του ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό ποσοστό οχημάτων τα οποία φτάνουν στο τέλο του κύκλου ζωή του, αλλά δεν ανακυκλώνονται ή αναχρησιμοποιούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή ε, τα οποία ενδεχομένω έχουν εξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρανόμω. Αυτή είναι λοιπόν η κύρια ανησυχία τη έκθεση και περιγράφει η τα οποια ενδεχομενω εχουν εξαχθει απο την ευρωπαικη ενωση παρανομω αυτη ειναι λοιπον η κυρια ανησυχια της εκθεσης και περιγραφει η εκθεση της προσπαθειας που καταβάλλονται και σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης, δηλαδή Επιτροπής Και γίνεται και λόγος και σε μια έκθεση η οποία θα συνοψίζει προηγούμενες εκθέσεις και η οποία θα είναι διαθέσιμη τον Αύγουστο. Με βάση λοιπόν εκείνη τη μελέτη του Αυγούστου θα ελπίζουμε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε περαιτέρω μέτρα τα οποία θα υποστηρίξουν τα όσα ήδη κάνουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα των απολεσθέντων εντό εισαγωγικών οχημάτων, των οχημάτων δηλαδή εκείνων που δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται. Θα ε, σταματήσω εδώ και βέβαια είμαι στη διάθεσή για να απαντήσω σε ερωτήματα. Σα ευχαριστούμε. Ο λόγο ε, τώρα στου συναδέλφου. Παρακαλώ. Κυρία Ντάλη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πιστεύω ότι κατ' ουσίαν ε, μιλάμε εδώ για το ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο η ζήτηση για τα αυτοκίνητα και έχουμε να κάνουμε με μια οδηγία που είναι καθοριστική σημασία όχι μόνο για τις οικονομίες μας αλλά και για το περιβάλλον. Και θεωρώ το όλο θέμα τόσο σημαντικό γιατί κατ' ουσίαν συνεπάγεται έρευνα για να εντοπιστεί η καλύτερη μεταχείριση των αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος ζωής τους, έτσι ώστε να υπάρχουν όσο δυνατόν και λιγότερα απόβλητα. Θα ήθελα να επισημάνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με περίπου 4,5 εκατομμύρια τέτοιου είδους αυτοκίνητα σε αιτήσια βάση. Ε, δεν ξέρουμε ε, τίποτα περισσότερο για αυτά. Μπορεί ε, να διαλύονται παράνομα, να υπάρχει παράνομη εξαγωγή τους. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή επισήμανε στην έκθεσή της για την εφαρμογή της οδηγίας της ότι ακόμα δεν έχει κατορθώσει να εντοπίσει αυτά τα αυτοκίνητα και κατά κάποιον τρόπο, ε, κατά την άποψή μου, η ίδια αμφισβητεί την εφαρμογή της οδηγίας. Και αυτά τα ε, αυτοκίνητα που κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται, ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να ρυθμιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ίσως να συστήσει μια ειδική ομάδα για να συντονίζει τη δουλειά στα κράτη-μέλη ή μήπως έχει κάτι άλλο κατά νου. Μήπως ε, να έχει σκεφτεί κάτι άλλο το οποίο ήδη εφαρμόζεται ε, να επιτρέπεται ένα είδος χρηματοδότησης, απόσυρσης που λέμε, για να ε, μπορούν και να διευκολύνεται η ε, δήλωση αυτών των αυτοκινήτων. Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά συνδέονται και με την ηλεκτρική κινητικότητα και τα ηλεκτροκινούμενα οχήματα. Εγώ σε τελική ανάλυση δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με την μπαταρία στο τέλος ε, του κύκλου της ε, ζωής ε, αυτών των αυτοκινήτων. Η μπαταρία που επιστρέφεται στην εταιρεία των αυτοκινήτων ή σε εκείνον που αναλαμβάνει να διαλύσει το αυτοκίνητο. Ο κ. Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, κοιτάξτε, η Επιτροπή εξετάζει θετικά την εφαρμογή της ε, οδηγίας ε, για... που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους. Τώρα, 4,5 εκατομμύρια είναι αυτά τα αυτοκίνητα κάθε χρόνο και δεν ξέρουμε πού καταλήγουν. Συμφωνώ με αυτά που μόλις τώρα ελέγχθησαν σχετικά με την ίχνη λασιμότητα, δηλαδή πρέπει να περιστεί στο ελάχιστο οι επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον, ε, τα διάφορα στοιχεία των αυτοκίνητων αυτών πρέπει είτε να ξαναχρησιμοποιηθούν είτε να ανακυκλωθούν. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα αυτοκίνητα και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για το περιβάλλον μας. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει αξιολογήσει τι πρέπει να κάνει για να εντοπίσει αυτά τα αυτοκίνητα. Και θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν και αρκετά νέα αυτοκίνητα τα οποία για διάφορους λόγους, κυρίως εμπορικούς, δεν ε, χρησιμοποιούνται ούτε βγαίνουν στην αγορά. Ε, κατ' ουσίαν γίνονται άχρηστα παρότι είναι καινούρια. Ε, η Κομισιόν τα έχει υπολογίσει αυτά και υπάρχουν άραγε κίνητρα για να χρησιμοποιηθούν τελικά τα αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν. Δεν είναι άχρηστα. άλλες παρακαλώ. Αν όχι, θα ήθελα να επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σωστά θέτεται το ζήτημα και αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της έκθεσης αυτής, δεν είναι καινούρια για τα οχήματα αυτά στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει με τις αρχές των χωρών μελών και πάντα ήταν πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη. Και το βλέπετε στις σελίδες 8 και 9 της έκθεσης κάποια παραδείγματα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μέτρα έχουν πάρει οι ίδιες οι χώρες μέλη για αυτά. Ένα από τα προβλήματα είναι η διευκόλυνση παράνομης επεξεργασίας των οχημάτων αυτών. Έχουν ληφθεί μέτρα όμως από τις χώρες για την αντιμετώπιση αυτών των ε, παράνομων ε, κέντρων ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις. Και αυτός βέβαια είναι ένας από τους... Ο τρόπος δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα είναι ακριβώς να ανοιχνεύσουμε αυτές τις παράνομες πρακτικές. Πρόκειται για μια σημαντική διάσταση. Άλλη σημαντική τώρα διάσταση είναι οι παράνομες εξαγωγές αποβλήτων καθώς εδώ υπάρχει το πρόβλημα του να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έχουν διαλυθεί ε, από τα οχήματα εκείνα τα οποία δεν έχουν διαλυθεί. Είναι δηλαδή, ε, θα πρέπει να δοθούν εδώ κατευθυντήρες γραμμές στις τελωνιακές αρχές προκειμένου να ε, λάβουν βοήθεια στις εργασίες τους. Επίσης, πριν από τρία χρόνια, τροποποιήθηκε ο κανονισμός για να επιτρέπονται πιο αυστηροί έλεγχοι από τις χώρες μέλη. Εγκρίναμε και έναν κατάλογο ε, συγκρισιμότητα, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε τους τελωνιακούς να αντιμετωπίζουν τις παράνομες εξαγωγές οχημάτων. Έχουν αναλυφθεί δηλαδή διάφορες πρωτοβουλίες μέχρι τώρα. Συγχρόνως, και το είπα λίγο, εκπονούμε μελέτη και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι, που εξετάζει όλες τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών μελών. Κάποιες αναφέρονται και στην έκθεση. Συγχρόνως θα δούμε τι παραπάνω μέτρα μπορούν να ληφθούν είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε επίπεδο χωρών μελών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σημαντικό ζήτημα των οχημάτων που χάνονται κάποια στιγμή, δεν μπορούν να βρεθούν με τίποτα. Κάποια στιγμή θα επανέλθουμε και θα συζητήσουμε τα πορίσματα της έκθεσης αυτής. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε με τις χώρες μέλη. Γιατί ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα μας επιτρέψει είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το πρόβλημα. Για την ερώτησή σας, τώρα, αν σας κατάλαβα, κατά πόσο η οδηγία θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως των εξελίξεων που έχουμε ηλεκτρικά οχήματα, μπαταρίες. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να συζητηθεί στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για τα απόβλητα, πρόταση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας ζήτησε να αναθεωρήσουμε και την οδηγία για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οπότε και αυτό είναι στο πρόγραμμα. Πράγματι είναι παλιά πια η οδηγία αυτή. Είναι το 2000. Οπότε θα ήταν λογικό κάποια στιγμή να αναθεωρηθεί. Ως Επιτροπή δεν έχουμε αποφασίσει πότε πρέπει να γίνει αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα πρέπει να ξαναδούμε εν ώψη μια τέτοια αναθεώρησης, μεταξύ άλλων αυτό που είπατε κι εσείς. Πάντως ήδη συζητιούνται διάφορε αναθεωρήσεις. Η οδηγία για τι μπαταρίε, για παράδειγμα, θα αναθεωρηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Οπότε, ίσω κάποια από τα θέματα για τις μπαταρίες που σας απασχολούν να λυθούν και στα πλαίσια της αναθεώρησης αυτής της οδηγίας για τις μπαταρίες. Έρχομαι τώρα στα νέα οχήματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για το ποια ακριβώ είναι η ερώτηση, αλλά έχουν υπάρξει email ανάμεσα ε, στο βοηθό σας για το θέμα αυτό. Τα νέα οχήματα μπορούν να γίνουν απόβλητα ή τα δοκιμαστικά οχήματα δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε ακριβώς. Πρόκειται για αυτοκίνητα τα οποία δεν βγαίνουν στην αγορά, δεν βγαίνουν καν, ε, διότι ε, προσπαθούν οι έμποροι να κρατήσουν ψηλά τις τιμές των αυτοκινήτων και τι γίνεται. Παράγονται τα αυτοκίνητα αλλά δεν βγαίνουν καν στην αγορά. Είναι αρκετά τώρα αυτά τα αυτοκίνητα και πρέπει να δούμε τι τα κάνουμε, να τα λάβουμε υπόψη μας. Ε, ίσως ε, ε, θα πρέπει κάπως να το εξετάσουμε περισσότερο το θέμα. Σας λέω και αυτά πρέπει να τα υπολογίζουμε γιατί εδώ δεν πρόκειται δεν ξέρει κανείς ε, πού θα καταλήξουν ε, αυτοί τα αυτοκίνητα. Ίσως και αυτά τα αυτοκίνητα να καταλήξουν ε, απόβλητα, να διαλυθούν και να χάσει κανείς κάθε ίχνος για το πού θα καταλήξουν. Τότε είναι και αυτό ένα παράδειγμα των οχημάτων που μπορεί να είναι καινούρια, αλλά που δεν περνάνε στην αγορά, άρα εξαφανίζονται, δεν καταγράφονται. Νομίζω ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των χαμένων οχημάτων. Βέβαια, κανονικά, εμείς μιλάμε για τα παλιά που χάνονται, έτσι. 3,5 με 4 εκατομμύρια είναι τα οχήματα που είναι πολύ πιο παλιά από αυτά που λέτε εσείς, που είναι στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Εσείς μιλάτε για μια διαφορετική κατηγορία. Πάντως αν έχετε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, τότε σας παρακαλώ να μας τη στείλετε. Εγώ είδα μια πολύ σύντομη ανταλλαγή mail μεταξύ νομίζω των βοηθών σας και των υπηρεσιών μου. Αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, ευχαρίστως να το εξετάσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και ολοκληρώνεται και η συνεδρίασή μας για σήμερα. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί στις 9 και αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Καλό βράδυ σε όλους.